So, ladies... Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο δεύτερο ήμιση της ε, συνεδρίασης της, ε, ΑΦΕΤ. Θέμα 13, έκθεση σχετικά με την έκθεση Επιτροπής του 2018 για τη Σερβία. Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι μας περιμένουν μερικές ψηφοφορίες και πάντοτε κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών μου ζητάει ο φίλος Κλίκεσταίν ε, να βιαστώ όσο γίνεται περισσότερο και ο φίλος κύριος Ζώστινιακ μου λέει ότι προχωράω με πάρα πολύ γοργούς ρυθμούς. Θα προσπαθήσω λοιπόν να ισορροπήσω ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα αλλά βεβαίως θα ακούω προσεκτικά αυτά που έχετε να μου πείτε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, μπορούμε αμέσως να περάσουμε στην ψηφοφορία. Για να δούμε, για να συγκεντρωθούμε όλοι. Συμβιβαστική πρόταση 1. Παρακαλώ. Σερβία, Σερβία. Μιλάμε για το 13, έκθεση της Επιτροπής για τη Σέρβια. Συμβιβαστική πρόταση 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6. Υπέρ κατά Μισό λεπτό, μισό λεπτό. 59, 59, κύριο Σόλτσα. Γιατί διακόπτεται τη διαδικασία. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία του κυρίου Σόλτ, Ποιο είναι κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84. Σαφχάουζερ, Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Κύριε Σαφχάουζερ, γιατί καταψηφίσατε την τροπολογία σας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ναι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για να δούμε. Πού πάμε τώρα. 186 ο κύριε Σαφάουζερ, υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 21 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, περνάμε συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Συμβιβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στο 227 φιλελεύθερη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.35 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.36 υπέρ κατά αποχές Α, μισό λεπτό να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε για το 236, τροπολογία 236, αρχίζει η ψηφοφορία. 56 συνάδελφοι ψήφισαν, τρει, τρεις φαντάζομαι ότι κοιμούνται, 58 παρόντες πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε 32 και 18 κατά. 228 υπέρ κατά αποχές. Για να το ελέγξουμε, το 200, το τροπολογία 228 αρχίζει η ψηφοφορία. Τέσσερις συνάδελφοι συνεχίζουν να μην συμμετέχουν. Μάλλον τρει συνάδελφοι υπέρ, Πέρασ ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 2.37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε και πάλι, ψηφίζουμε για την τροπολογία 237. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. να δούμε όλες αυτές τις ιδεολογικές εκθέσεις. 17 ως 21 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 για να ελέγξουμε. 27 Για να ελέγξουμε την 26, αρχίζει η ψηφοφορία των ε, Ντέλη και Μπόσκορ. Μπόσκορ. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε 43 με 5. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 28 υπέρ, 28, 28 υπέρ, κατά, αποχές για να ελέγξουμε για την 28, ο του κύριου Σόλτ. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 33 και 34 υπέρ, κατά, αποχές. Για να το ελέγξουμε, ελέγχουμε 33-34 τις απολογίες, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Περνάμε στα εκτιμώντας, υπέ, ένα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έξι με 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11-12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα ότι απορρίπτεται, αλλά για σιγουριά να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Vote Πέρας ψηφοφορίας ε, εγκρίθηκε. Τέλος, 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για όλη την έκθεση, σχέδιο έκθεσης. Μας λείπει ένας. Πέραση της εγκρίθηκε 49 υπέρ 3 κατά συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε τώρα στο 14. Έκθεση σχετικά με την έκθεση τη Επιτροπής του 2018 για το κοσυφοπαίδιο. Ο εισηγητής θα ήθελε να πάρει το λόγο, όχι. Προχωράμε λοιπόν. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Doing Anders. Fine, and you? How's your kid? Fine. Close. The vote is closed. It's been rejected. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται.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 Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 του κυρίου Σαφόζερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «187» του κυρίου Ζόρνιας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 195 αντάκτουσον. Είναι ακόμα μέλος του Κοινοβουλίου. Είναι βουλευτής στη Σουηδία τώρα. Ποιος είναι υπέρ του Σουηδικού Κοινοβουλίου, υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. 195 άρχεται η ψηφοφορία. Five colleagues missing. Πέντε συνάδελφοι λείπουνε. Αντάκτουσον is missing. <laughs> so. Ο Αντάκτουσον λείπει. Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 208 Μίλαν Μόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 231 αντάκτουσον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 232 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 234 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 235 υπέρ κατά αποχές. 235 ηλεκτρονική επαλήθευση του κυρίου Μίλαν Μόν. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 30 ψηφί υπέρ 20 κατά. Recitals. Number 10. In favor. Αιτιολογικές σκέψεις 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 12 και 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται, 14 υπέρ κατά αποχές εγκρι... απορρίπτεται, 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στη 18 πάμε, Σαφόζερ υπέρ κατά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 Πέρα τη ψηφοφορία. 37 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Φτάνουμε σε αιτιολογικές αναφορές. 1. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της 8. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 31 ψήφοι υπέρ, 20 κατά. 9 υπέρ, κατά αποχές. Οι φιλελεύθεροι καταψήφισαν πριν η ηλεκτρονική επαλήθευση και τις 9. have the liberals, you can see. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28 υπέρ, 24 κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία πάνω στο σχέδιο ψηφίσματος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Two colleagues what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 Αποχές. Ας επιβεβαιώσουμε. Άρχεται η ψηφορία. Λίγη. Υιοθετήθηκε 29 εναντίον 27. 17. Του κ. Κούκαν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παρα... Ε, τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Κ. Κόβατσεφ ξανά υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμόν 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Καστάλτο υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Door is Λίγη. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική προθεμόν 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύουμε. Vote is open.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 34 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. 69 κατά πίπτη. 70 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται έτσι δεν είναι. Επαληθεύουμε την 70. Εγκρίνεται. 32 υπέρ 23 κατά. Συμβαστική 14 υπέρ κατά Αποχέ, εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά Αποχέ, απορρίπτεται. Συμβαστική παρθμό 15 υπέρ κατά Αποχέ, εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές. Επαληθεύουμε την 83. Closed. Λήξη ψηφοφορία εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 89. Δύο τμήματα. Με έτοιμα του κ. Πίτσουλα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε το πρώτο τμήμα της 89. It's closed. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Closed. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. Ε. Ωραία. Επαληθεύουμε την 96. Close. 28 υπέρ 27 κατά. Εγκρίνεται. 95 του κ. Χατζηγεωργίου υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 107. Ανδρουλάκης και Μάρτιν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 111 υπέρ, κα... Το κ. Καστάλτο είναι. 110 ζητάτε επαλήθευση. Ξεκινάει η ψηφοφορία ότι είναι 110. 110 the vote closed. Λίγη ψηφοφορία, εγκρίνεται 49 υπέρ από τα κατά. 111. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. Ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά, εποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, εποχέ εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά, εποχέ. Επαληθεύουμε την 118. Εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε ξανά. 119 του κ. Μέζεριτς. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε την 129. Against, but we better check. It's closed. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 134 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 135 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 136 κατά πίπτη. 137 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 138. 139-140 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτονται, απορρίπτονται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική έκθεση. Παράγραφος παριθμών 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία παραθυμών 1 και 2 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, απορρίπτονται Επαληθεύουμε. Ναι. Τροπολογίες 1 και 2. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαρθμών 5 υπέρ κατά αποχές. Επαληθεύουμε την 5. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου, όπως τροποποιήθηκε, άρχεται η ψηφοφορία. Δεν έχουν ψηφίσει δύο συνάδελφοι. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 47 ψήφοι υπέρ, 5 κατά. Συγχαρητήρια κύριε Τάνοκ. Περνάμε στο σημείο 16. Έκθεση της Επιτροπής για την πρώην Οικοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο κ. Βάγκελ θέλει το λόγο. Δεν έχω τίποτα κύριε Πρόεδρε. Μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε με την τροπολογία 31 της κυρίας Σακοράφα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 σε Ψήφι υπέρ κατά αποχές. Για να το ελέγξουμε. Αλλά νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Τέλος ψηφοφορίας. 27 τα 26 απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60. κυρίω αυχάζω. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 Καστάλτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 Κύριε Βίστησεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές. Για να ελέγξουμε, ελέγχουμε την 80. Τροπολογία 80. Τελείωσε η ψηφοφορία, απορρίφθηκε. 81, τζαμπάσκι, υπέρ, κατά, αποχές τι σήκωσε κανένα στο χέρι του 81 αρχίζει η ψηφοφορία Επτά συνάδελφοι μας λείπουν. Έξι συνάδελφοι, πέντε, τέσσερις. Ωραία, τελείωσε η ψηφοφορία. 39 υπέρ 8 κατά εγκρίνεται. Περνάμε μετά 8 ε, ε, υπέρ κατά 83 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε του κυρίου Πίκουλα υπέρ κατά με ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 26, 25 υπέρ, 25. Συμβαστική 8 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται, 93 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 92 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 91 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 κούμπατσεπ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για να ελέγξουμε την 98. Η πιο σημαντική ψηλοψηφοφορία, Αντρέα, στην πολιτική σου καριέρα είναι αυτή. Μας λείπουν τρεις. Συνεχίζουν να λείπουν τρεις. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε αυτό. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 Καστάλντο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 κυρίε αγοράφα υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την 115. 115. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε 28 υπέρ, 26 κατά, συμβαστική 12 υπέρ κατά και 90, 23, 123 καστάλτο εγκρίνεται, Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται 131 μέζερες υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 132 μέζερες υπέρ κατά αποχές. Για να το ελέγξουμε, ελέγχουμε την 132, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Εγκρίθηκε. Πού είμαστε? 133. Καστάλτο Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να το ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 133. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Νταμπάτσικη. 134. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές για να ελέγχουμε ελέγχουμε την 136 τη της απορρίφθηκε Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 137 υπέρ κατά εγκρίνεται, λιγοτό, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 τσαμπάσκι υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 159 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας σαφώς έχει αγριθεί, 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 161 υπέρ κατά απορρίφθηκε 162 υπερκατά απορρίπτεται 162 υπερκατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές 165 για να το ελέγξουμε αρχής ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 166-67 ε, υπέρ κατά για να ελέγξουμε 167 ψηφίζουμε πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε 168 πώς υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά 179 ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 17 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 18, ε, 196 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την 196 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απολύφθηκε. Εκατόν ενενήντα πώς υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε 197 Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 212 σε πρώτο δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.14 κούκανε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2.15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 2.16 υπέρ κατά τα αποχές εγκρίνεται. 2, 17, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2, 19 υπέρ κα, καταπίπτει. Ευτυχώς. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2, 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην αιτιολογική έκθεση. 1 ε, υπερκατά, δύο ε, ε, ε, ε, ε Εγκρίνεται. Περνάμε στο 17 υπέρ αιτιολογική έκθεση. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 18 υπέρ απορρίπτεται, 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 20 υπέρκατα κατά αποχές απορρίπτεται, 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε το 23 αρχίζει η ψηφοφορία πέραση ψηφοφορίας σαφώς εγκρίθηκε 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όλη η τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. τριάντα 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η αναφορά, 2 υπέρ, υπέρ, κατά, α, για να το ελέγξουμε, είμαστε στην αιτιολογική αναφορά. Δύο, ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Α, καταπίπτει η ένα, η τρία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, αιτιολογική αναφορά πέντε υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται, έξι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για να, ελέγχουμε, ε, να ελέγξουμε αιτιολογική αναφορά 6. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 28-27. 7 αιτιολογική αναφορά, 7 υπερκατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχίζει η ψηφοφορία για όλη, όλο το σχέδιο έκθεσης. Τρεις συνάδελφοι λείπουν, δύο συνάδελφοι λείπουν, ένας συνάδελφος λείπουν. Μα κάποιος κοιμήθηκε εδώ, υπάρχει ένας που δεν συμμετέχει σε καμία ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας, 47 υπέρ, 9 κατά, συγχαρητήρια, περνάμε τώρα. Στην επόμενη ψηφοφορία, έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την Αλβανία. Μήπως θα ήθελε ο Κνούτ Φλέκενστάιν να πάρει το λόγο. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. 57 επαλήθευση, ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Oh, this has been rejected. Πέρα στις ψηφοφορίες απορρίπτεται. Ωραία. 58 υπέρ. Κατά άποχες. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση. Ωραία. 60. Άρχεται η ψηφοφορία. The τη ψηφοφορία closed. ψηφοφορίας. 50 κατά, 4 υπέρ. Επαληθεύσαμε και περνάμε στη συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 67 Καστάλτο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 94 κούκαν υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 98 σωράγια πόστη υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση της 98 άρχεται η ψηφοφορία. Closed. This has been rejected. Απορρίπτεται. 100, Mr. 100 Ζόσνιες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 101 και 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 103 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση της 104. Άρχεται η ψηφοφορία. It's τη Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές... 113 ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα closed. Πέρας απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση της 122 Helmut Scholz. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση της 128. Άρχεται η ψηφοφορία. Ναι, είναι αρκετά σαφές. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία 129. It's closed. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση και της 130. 1-3-0. τη εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 132. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Σαφώς εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 165 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 166 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Εγκρίθηκε. 167 ε? υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, σκέψεις 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 του κυρίου Κουκκαν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ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 The vote is now closed. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεμε 44 ψήφους υπέρ, 5 ψήφους κατά. Συγχαρητήρια στον κύριο Συγητή. So we have another very long voting list. Έχουμε άλλη, άλλο ένα κατάλογο αρκετά μακροσκελή με πολλές συμβαστικές προτάσεις. Απίστευτο. Συμβαστική υπαριθμόν 1 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την έκθεση για τη Γεωργία, έτσι το ξέχασα να σας το πω. τριάντα 31. Κύριε Τάνοκ, υπέρ του κυρίου Τάνοκ, συγγνώμη, υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Όχι. 46 μαμίκινς. Μαμίκινς. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 έχει αποσυρθεί ευτυχώς. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5-57 έχουν αποσυρθεί. 60 μαμίκης υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 74. Α, αποσύρθηκε. Ευχαριστούμε κύριε Γιούρεκ. Μπράβο. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 97. Τη κυρία Χάρμ. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Επαληθεύουμε. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 106. Το αντιπρόεδρο. υπέρ. Α, συγγνώμη. Βιάστηκα. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην 106. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές. Επαληθεύουμε την 109. Vote is closed. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. 140 του κ. Σόλτς υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση για τα 141. Εγκρίνεται. 143 του κ. Καστάλτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τη κυρία Χάρμς 144 υπέρ κατά αποχέ. απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχέ. επαληθεύουμε τη συμβιβαστική 17. Right, the vote is closed. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 21 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 95. Τι σχέση έχει η με εμά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλο πάντων, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 24, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Είναι τα 14, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 25, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 219, υπέρ, κατά, αποχέ. Εγκρίνεται. 2.20 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 2.21 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Είναι τα 7 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 2.22 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 3 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 2.24 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 16 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 2.25 έχει αποσυρθεί. Είναι τα 15 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται.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 Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ten colleagues missing. Wake up. Δέκα συνάδελφοι κοιμούνται. Ξυπνήστε. Επτά, πέντε μένουν ακόμα, τέσσερις. Λίγη ψηφοφορία. 43 υπέρ, 7, 7 ε, κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια στον κύριο Μαμίκιντς. Έκθεση για τη Συμφωνία Σύνδεσης με τη Μολδαβία. Ο κύριος Αουστερβίτσιος θέλει το λόγο. Ο, ζήτω Μολδαβία. Ζήτω Μολδαβία, ζήτω και εμείς.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 εποχές. Επαληθεύουμε την 65. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77. Αστροβίτσιος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 106 της κυρίας Νικολά υπέρ. Κατά αποχές. Την επαληθεύουμε. 106 επαληθεύουμε. The vote is closed. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. 12 συγγνώμη. Για την παράφου 13. Υπέρ. Κατά αποχές επαληθεύουμε. Συμβαστική υπαριθμών 12. εγκρίνεται. 35 υπέρ, 17 κατά. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά, αποχέ. απορρίπτεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, απόχε. επαληθεύουμε την 14, συμβαστική πρόταση 14. The vote is closed. Εγκρίνεται. Τροπολογία 165, Σαφχάουζερ, υπέρ. Κατά, αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15, υπέρ. Κατά, αποχέ. Επαληθεύουμε τη 15. Compromise 15. The vote is open. The vote is closed. 48 to 2. 48 υπέρ 2 κατά. Περνάμε στην ίντα 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 181 ε, Στρεβίτσιους υπέρ κατά εποχέ. εγκρίνεται 182 υπέρ κατά εποχέ. εγκρίνεται 57 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται 57 υπέρ κατά εποχέ. εγκρι... ε, ε παληθεύουμε Ναι. Εγκρίνεται. 6. έκθεση. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 6. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 7. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. τα 3. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2. Υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται. Είναι τα 5 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται. Είναι τα 6 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται. επαληθεύουμε τη 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. εποχέ. Επαληθεύουμε τη 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Υπαριθμόν 1 αναφορές ε, υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε την αναφορά υπαριθμών 1. 2 υπέρ. Κατά. εποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 31 ψήφοι υπέρ, 5 κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ο Θεός να το φυλάει. Περνάμε στη δεύτερη μεγάλη ψηφοφορία. Περνάμε στο 20 ενδιάμενη έκθεση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 21-27 η θέση του Κοινοβουλίου εν ώψη συμφωνία. Η συγγήτρια συντάκτρια νομοθότησα Μαρίκε Η κυρία Σάκη είναι εδώ παρούσα, όχι. Οπότε δεν μπορεί να μας πει και τίποτα. Περνάμε στον ε, κατάλογο της ψηφοφορίας. Συμβαστική πρόταση 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές. Για να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 13 το πρώτο μέρος. Τροπολογία 13 το πρώτο μέρος. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τροπολογία 13, δεύτερο μέρος, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3, υπέρ κατά εγκρίνεται υπέρ κατά εγκρίνεται 26 γιώτης ψήφι υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την 26 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε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 Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε την 32 αρχή της ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 33. Ε, Γιώργη Σολέ υπέρ. Κατά. Αποχές για να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για την 33. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Περνάμε στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, σχέδιο γνωμοδότησης. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 35 υπέρ, 4 κατά, 11 αποχές. Ή το αντίθετο. Dear colleagues, it's the last... Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στην τελευταία σημερινή μας ψηφοφορία. Μερικέ Μερικές από αυτές τις τροπολογίες αποτελούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 35 υπέρ. Κατά αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας πληροφορίας. 21-20. Ωραία, καλή είδηση για τον κύριο Κίλαμ. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά. Για να δούμε. Εγκρίθηκε. Για να το ελέγξουμε. 47. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 50 υπέρ κατά αποχές για να το ελέγξουμε 50 αρχίζει η ψηφοφορία Ψηφίζουμε για το 50. 50. Πέρας ψηφοφορία εγκρίθηκε. Κατάλαβα καλά ότι ο κύριος Φλέκενστάιν θέλει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 49. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, για το ελέγξουμε 59, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 60 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές. Για να ελέγξουμε το, την τροπολογία 61. Αρχίζει η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, 67 υπέρ κατά αποχέ. Για να ελέγξουμε. 67 Βαλέρο. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 4 υπέρ κατά τα ποχέ εγκρίνεται, 77 υπέρ κατά ποχέ εγκρίνεται, 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 συμβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται, 82 υπέρ κατά αποχές, το ελέγχουμε, αρχή της υποφορία, 82, την 82, πέρας ψηφοφορίας, απορρίφθηκε. 83 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές για να το ελέγξουμε ελέγχουμε την 86 86 Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 90. Ζαμπίνα Λούζινγκ υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 103 υπέρ κατά αποχές, για να ελέγξουμε το 103, τροπολογία 103, πέρας ψηφοφορίας, από ό,τι φαίνεται εγκρίθηκε. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε την 108 The vote is Πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να δούμε τι αυτό. Δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Για να ελέγξουμε την 109. αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές. Για να ελέγξουμε το 111. Πέρας. Εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 καταπίπτει 115 καταπίπτει 117 καταπίπτει 118 ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική πρόταση 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 130. Τα υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 149 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές για να ελέγξουμε για να ελέγξουμε Υπέρες πληροφορίες εγκρίθηκε 154 βανόνται, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Αιτιολογική έκθεση 6 υπέρ κατά ε, ποιες εγκρίνεται, 7 υπέρ κατά ποιες απορρίπτεται, η 9 ε, υπέρ κατά ποιες απορρίπτεται, 8 αιτιολογική έκθεση υπέρ κατά ποιες απορρίπτεται, 10 υπέρ κατά ποιες απορρίπτεται, 11 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όλες αυτές οι τροπολογίες είναι στην αιτιολογία έκθεση. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 18 υπέρ κατά αποχές, για να ελέγξουμε την, ε, τη λογική έκθεση 18, αρχίζει η ψηφοφορία. Τελείωσε η ψηφοφορία, απορρίφθηκε. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 20 υπέρ, κατά, αποχές, για να ελέγξουμε το 20, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας,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 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Α, τι για την 31 δεν ψηφίζουμε. 32 ε, παρνιό υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές εμπορύπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές. Για να ελέγξουμε 34, αρχίζει η ψηφοφορία.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 Λείπουν οκτώ συνάδελφοι. Παρακαλώ. Αποχές. Αποχή. Πέντε συνάδελφοι λείπουν. Σας παρακαλώ. Ωραία πέρας πιοφορίας. 27 ε, υπέρ, 12 κατά, τέσσερις αποχές, διάλειμμα ένα λεπτό και περνάμε στο 22 μετά της μερισίας διάταξης. Συνάδελφοι, πρέπει να συνεχίσουμε. Φτάνουμε στο σημείο 22. Ενημέρωση σχετικά με την αποστολή της Επιτροπής ΑΦΕΤ στο Καζακστάν και στο Ουσπεκιστάν 17 με 21 Σεπτεμβρίου 2018. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πραγματοποίησε αποστολή στην Αστάνα, στο Καζακστάν δηλαδή, και στο Ουσπερκιστάν, στη Σαμαρκάντη και στην τασκεντη 17 με 21 Σεπτεμβρίου, για να διευρυνθεί ο πολιτικός διάλογος και η κυροβουλευτική διάσταση και η, την, απο, της αποστολής ηγήθηκε ο κύριος Κρίστιαν Πρέντα. Έχει το λόγο, Κρίστιαν, παρακαλώ. Ε, voilà. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, δημιουργήσαμε μια επίσκεψη στο Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν ως ΑΦΕΤ. Δύο, χώρες στο, δύο μέρες στο Καζακστάν, δύο μέρες στο Ουσμπεκιστάν. Ο γενικός στόχος ήταν με τους συνομιλητές μας να ανταλλάξουμε απόψεις για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Κεντρική Ασία. Πολλές από τις συναντήσεις ήταν εξαιρετικά χρήσιμες. Συναντήσαμε για παράδειγμα στο Καζακστάν τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, ο οποίος μας αφιέρωσε πολύ χρόνο. Συναντηθήκαμε επίσης με τα μέλη της Επιτροπής Διεθνών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Άμυνας και της Ασφάλειας Πολλά από τα μέλη της Επιτροπής αυτής ήταν παρόντα και ο πρόεδρος βέβαια. Και κατά τη διάρκεια αυτών των ανταλλαγών, όπως και κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την Συνταγματική Επιτροπή του γερουσίας. θίξαμε ένα αριθμό σημαντικών θεμάτων που άπτονται των σχέσεων Καζακστάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίση στήξαμε και το θέμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έγινε διάλογος, θερμός, Μερικές φορές χρειάστηκε να εξηγήσουμε καλύτερα τις θέσεις μας, γιατί ε, αυτοί δεν καταλάβαιναν πολύ καλά τη σύνδεση ανάμεσα στις εξωτερικές υποθέσεις και τα δικαιώματα του ανθρώπου. συχνά οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν βλέπουν αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στα δικαιώματα του ανθρώπου και τι εξωτερικέ υποθέσει. Αυτό είναι ένα φαινόμενο αρκετά κοινό. Οπότε χρειάστηκε και εμεί να είμαστε λίγο διδακτικοί. για να διευκρινίσουμε την άποψή μας. Είχαμε δύο αρκετά διαφορετικές εμπειρίες μεταξύ Αστάνα και Αλμάτι. Η, Αλμάτι ε, η μητέρα ενός κατάδικου φυλακισμένου ε, ήρθε να μας δει και βγαίνοντας από το ξενοδοχείο τη συλλάβανε και δεν ξέρουμε πού την πήγαν. Ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο. Ευτυχώ η πρέσβης του Καζακστάν στις Βρυξέλλε ήταν εκεί δίπλα και ζητήσαμε τη βοήθειά της. Μα είπαν κάποια στιγμή ότι αργότερα ότι απελευθερώθηκε. Αλλά αυτό μας υποχρέωσε να ακυρώσουμε μια συνάντηση και μας φόβησε κιόλας λίγο. Γιατί αμέσως μετά είχαμε να δούμε τους εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και οι ιστορίες τους είναι πολύ δυσάρεστες, πολύ σοβαρές. Οπότε το ερώτημα είναι μπορεί να γίνει ειλικρινής διάλογος με τους φίλους από το Καζακστάν. Προσπαθήσαμε να θίξουμε και τα ενεργειακά και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και υπό την οπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δύσκολο αυτό. Ε, χρειάζεται προσπάθεια. Έχουμε και την επίσκεψη Παντζέρη και πολύ καλά που είναι εδώ, διότι ο κ. Παντζέρη θα επισκεφθεί το Καζακστάν ως πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, θίξαμε αυτή την επίσκεψη, τον περιμένουν, οπότε ζητήσαμε να επισκεφθεί τους ανθρώπους για τους οποίους μιλήσαμε με τους συνομιλητές μας, τις φυλακές, να, να επισκεφθεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν φυλακιστεί εξαιτία της δράσης τους υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι θα, θα είναι εφικτό και ότι θα έχει πρακτικά αποτελέσματα με απελευθερώσεις ανθρώπων για τους οποίους μιλάμε εδώ και πολύ καιρό. Θίξαμε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ο αναπληρωτής Γενικός Αγγελέας μας δέχτηκε του αναφέραμε συγκεκριμένα ονόματα, μας έδωσε πληροφορίες, είπε ότι είναι πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί μας. Αυτή την καλή θέληση την είδαμε και στη Βουλή. Οπότε ελπίζουμε ότι η επίσκεψη Παντζέρη θα είναι ευκαιρία για να εμβαθυνθεί ο διάλογος για την προστασία των ελευθεριών. Σας είπα στην αρχή ότι συναντήσαμε ένα αριθμό καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Ναζαρμπάιεφ στην Αστάνα. Ε, πρόκειται για Ευρωπαίους και Αμερικανούς υπηκόους που βρίσκονται εκεί, στο πλαίσιο ενό εκπαιδευτικού συστήματο, το οποίο από ό,τι μα είπαν είναι ψηλή ποιότητα και δεν ελέγχεται από το κράτο. Έχουμε πανεπιστήμιο της, των ΗΠΑ, της Σιγκαπούρης κλπ. που έχουν φτάσει στο Καζακστάν και διδάσκουν χωρίς να ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα, δύο λόγια για το δεύτερο σκέλος της επισκεψής μας. Σκένδη και Σαμαρκάνδη. Εκεί συναντηθήκαμε με την κοινωνία των πολιτών. Ορισμένοι από αυτούς αμφισβήτησαν τις επίσημες τοποθετήσεις, την επίσημη θέση ότι έχουν απελευθερωθεί όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Εμείς προσπαθήσαμε, συναντώμενοι με τους αξιωματικούς αξιωματούχους, να διαπιστώσουν ποια είναι η αλήθεια. Η Άννα Γκόμες ήταν εκεί, στην Τανσκένδη, είδαμε ότι οι συνομιλητές μας έδειξαν μια, ένα ανοιχτό πνεύμα και το Κοινοβούλιο και το Υπουργείο Εξωτερικών επιθυμούν να επωφελθούν τη ευκαιρία. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή το Ουσμπεκιστάν περνάει μια διαδικασία ανοίγματο και α, ανταγωνίζεται σε αυτό το θέμα με το Καζακστάν. Έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα θέματα τα οποία τρέχουν. Για παράδειγμα, σχετικά με το Αφγανιστάν και το πώς οι Ουσμπέκοι μπορούν να βοηθήσουν στις διαπραγματεύσεις εκεί. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών στο Αφγανιστάν για να δούμε ποιο θα είναι το καινούριο πανόραμα. Επίσης συζητήσαμε εκεί με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων που βρίσκονται εκεί για θέματα εγκληματικότητας, ε, εμπορίων ναρκωτικών, προληπτικής διπλωματίας, πολύ σημαντικό και αυτό. Και είχαμε και την ευκαιρία με τους Ουσμπέκους συνομιλητές μας να ανταλλάξουμε πολλές ιδέες για το σύνολο της Κεντρικής Ασίας. Και για το πώς βλέπουν αυτή την Ευρώπη. Μετά στη Σαμαρκάνδη συζητήσαμε με τις ε, περιφερειακές αρχές τον ε, αναπληρωτή του κυβερνήτη και εκεί συζητήσαμε για δύο θέματα. Καταρχήν ένα σχέδιο που έχει σχέση με την προστασία των γυναικών έναντι οικιακής βίας, το οποίο ήδη εφαρμόζεται, υλοποιείται, και ένα άλλο σχέδιο για την διαχείριση τεραιών αποβλήτων, το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία. Εκεί είδαμε ένα κάποιο ενδιαφέρον και οι δύο χώρες, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν, συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό για θέματα εξωτερικής πολιτικής Συζήτησαμε τη Συρία, ε, τη συνθήκη μη διάδοσης, τη μη διάδοση γενικά. Και οι δύο πλευρές, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν, μας δήλωσαν ότι επιθυμούν και στο μέλλον να συνεχίσουν τη συνεργασία μαζί μας. Λυπάμαι κύριε, που κύριε Βέτα Κρικούλ δεν είναι μαζί μας, γιατί είναι η πρόεδρος της αντιπροσωπείας για, τη σχέση με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Ήταν μαζί μας στο πρώτο κομμάτι, στο πρώτο σκέλος της επισκεψής μας, στο Καζακστάν. Και είναι σημαντικό όχι απλώς να συνδέουμε τη δουλειά μας με την αντιπροσωπεία της χώρες της Κεντρικής Ασίας, αλλά και μεταξύ μας συνδέομαστε Κάποιος μας είπε επί τόπου ότι δεν μιλάμε ποτέ για ανθρώπινα δικαιώματα όταν πάμε επί τόπου. Αυτό είναι ανησυχητικό. Οι αντιπροσωπείες όταν βρίσκονται στο εξωτερικό δεν μπορούν να δρουν ως ομάδες φιλίας. Θα πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, Κριτιάν, για την ενημέρωση. Από ό,τι γνωρίζω, η κυρία Αναγκόμε. πήρε μέρο σε αυτή την αποστολή, οπότε κυρία Γκόμε, έχετε το λόγο. Συμφωνώ με όσα ήδη υπόθηκαν από τον Κρίστιαν. Εγώ θα ήθελα να σας πω την προσωπική μου άποψη είδαμε δύο χώρες που ακολουθούν μία εντελώς διαφορετική πορεία. Το Καζακστάν ακολουθεί την ε, παλιά πορεία και βρίσκεται αντιμέτωπο με μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό είναι κάτι που μας είπαν, κάτι δίαν πάρα πολύ, όχι σε δημόσιες συναντήσεις, γιατί ε, τι να κάνουμε, έχουμε να μπροστά μας ε, ε, ε, ε, μία, με μία δικτατορία. Εγώ μπορώ να το συγκρίνω με την εποχή που στην Συρία ήταν επικεφαλής ο πατέρας του Ασάντ. Από την άλλη πλευρά συναντάει κανείς πολύ ενδιαφέροντες, πολύ καλλιεργημένους ανθρώπους και δίχως άλλο η προσέγγιση τους ήταν πολύ ανοιχτή, πολύ εξωστρεφής. Ο Ξίστα αναφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο. Ναι, θα, θα ε, ε, συναντούσα δέκα καθηγητές οι οποίοι αμείβονται από αυτό το πανεπιστήμιο, είναι ξένοι, καταλαβαίνετε ότι δεν θέλεγαν κατά του πανεπιστημίου, ε, πληρώνονται, πληρώνονται για να είναι εκεί και να μιλάνε καλά. Και συναντήσαμε και έναν φοιτητή. Ένα φοιτητή. Ε, όταν πηγαίνει κανεί σε ένα πανεπιστήμιο μια οποιασδήποτε άλλη χώρα, δεν περιμένει να βρεθεί αντιμέτωπο με κάτι τέτοιο. Μίλησα με αρκετού ανθρώπου και πραγματικά ανησυχούν γιατί είναι 77 ετών ο ηγέτης του Αζερβαϊτζάν και πολλοί φοβούνται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το μέλλον. Και πραγματικά φοβούνται ότι τα πράγματα θα είναι μάλλον πολύπλοκα στο μέλλον. Υπάρχει ε, και ένα υφέρπον εθνικισμός ε, αυτό είναι κάτι που δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Πήγα στην Αλμάτη, στην άλματι νιώσαμε, μόλον ότι δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες να καταλάβουμε, είχαμε την ευκαιρία να νιώσουμε ότι ήμασταν σε μία πραγματική πόλη. Μιλάμε ε, για μια τεχνητή πόλη που υπάρχουν κτίρια, που μεγάλα, δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι, πολύ εντυπωσιακοί, αλλά όχι κατανάγκη. Ε, ευχάριστη. Ήταν σαφές ότι ο Υπουργός Εξωτερικών προσπαθούσε να προβάλλει μια συγκεκριμένη εικόνα. Στο μάτι όμως η εντύπωση ήταν ότι βρισκόμαστε σε μια πραγματική πόλη και εκεί αρχίζουν τα πράγματα να περιπλέκονται γιατί έγινε αυτό το συμβάν το οποίο αναφέρθηκε ο Κριστιαν και που είχε συγκεκριμένες επιπτώσεις για μας. Θέσαμε ερωτήματα για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πραγματικά όπως είπε και ο Κρίστιαν δεν ήταν αποδεκτό να μην θέσει ερωτήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς αναφερθήκαμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και πολύ καλά κάναμε. Έχουμε όμως την εντύπωση ότι δεν υπάρχει ελευθερία σε αυτή τη χώρα και οι άνθρωποι που ήθελαν να μας προσεγγίσουν δεν τα κατάφεραν, τους εμπόδιζαν. Ο είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη που θα κάνει ο Αντώνιο και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Αντώνιο να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα του δοθούν. Πάρα πολύ σημαντικό να πάει να μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ουσβεκιστάν, μισό λεπτό να τελειώσω. Μάνα, Άννα, σε παρακαλώ, πιέζει ο χρόνος. Πόσο θες να μιλήσεις ακόμα. Καλά, να μην μιλήσω, να σταματήσω. Συγγνώμη, όταν επισκέπτομαι ένα μέρος και πρέπει να σας ενημερώσω, δώστε μου λίγο χρόνο, αν δεν θέλετε, να μην μιλήσω. Όχι, όχι. Ε, ε, σε παρακαλώ, σύντομα. Πήγα στον Ουμπεσχιστάν πριν από αρκετά χρόνια, το 2012 και πραγματικά υπήρχε διαφορά. Υπάρχει ένα πολιτικό άνοιγμα τώρα. Πολλά από τα προβλήματα που θέσαμε και την αρχή, το θέμα της ε, εργασίας ε, ανηλίκων για παράδειγμα, έχει αντιμετωπιστεί. Και αυτό αρκετά ακριβώς ε, αυτή την ιδέα μας μετέφερε η κοινωνία των πολιτών Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ξεχαστεί στις φυλακές για διάφορους λόγους, αλλά η κοινωνία των πολιτών είχε τη δυνατότητα να μας προσεγγίσει, πράγμα που δεν έγινε στο Καζακστάν. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μία σχέση με το Καζακστάν για θέματα ενέργεια, οτιδήποτε άλλο και καταλαβαίνω ότι είναι μία χώρα στρατηγική σημασία. Βέβαια, δεν πρέπει να παραμελούμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλουμε μια υγιή ε, ε, ε, ε σχέση, θα πρέπει, να πάψουμε ποτέ να τονίζουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι ώστε οι άνθρωποι που κυκλοφορούν με τα μπλε παλόνια να μην θεωρούνται ότι ε, ε, είναι ε, ανατρεπτική. Ευχαριστώ, άναγκό μας. Κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριος Σάφας έφυγε. Παρακαλώ, κύριος Μπούχνερ. Για την αποστολή ή για ποιο σημείο να σας μιλήσω. Α, για την αποστολή, ναι. Ήθελα πολύ σύντομα να προσθέσω ε, κάτι στα τελευταία λόγια της κυρίας Γκόμες. Έχω επαφές με πολίτες στο Ουσπεκιστάν. Προς τα έξω δίδεται η εντύπωση ως αν η χώρα να είναι πιο ανοιχτή, ενώ ε, στο εσωτερικό της χώρας πολύ λίγα έχουν αλλάξει. Για παράδειγμα, έχει καταργηθεί η παιδική εργασία κατόπιν πίεσης από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είπαμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε συμφωνία μπορεί για το μαμβάκι εάν αυτό παράγεται με παιδική εργασία. Και τι γίνεται τώρα, έχουμε καταναγκαστική εργασία των ε, ενηλίκων ε, αντί για των παιδιών. Επίσης έχουμε πολιτικούς κρατούμενους. Εγώ ήμουνα πρόσφατα εκεί και ήμασταν πολύ ενθουσιώδης για το πώς έχει ανοίξει η χώρα προς τα έξω, αλλά απομένουν πάρα πολλά να γίνουν ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπίχνερ για την παρατήρηση σας αυτή. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Από ό,τι βλέπω όχι περνάμε στο σημείο 23 της ημερησίας διάταξης. Έχουμε καθυστερήσει κατά μισή ώρα ή ίσως μπορέσουμε τώρα να επιταχύνουμε. Συνάδελφοι, φτάνουμε στο σημείο 23 της ημερησίας διάταξης, ετήσια έκθεση ε, σχετικά με την εφαρμογή της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Κάποιες παρατήρησεις από τη δική μου πλευρά διότι είμαι εγώ Η Εισηγητής είναι πάντα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Το σχέδιο έκθεσης μοιράστηκε πριν κάποιες εβδομάδες. Ελπίζω όλοι να είχατε χρόνο να την εξετάσετε πιο προσεκτικά. Ακόμα και, περισσότερο από την προηγούμενη ετήσια έκθεσή μου, ε, επέλεξα να εστιάσω στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της. Ε, η έκθεση ξεκινάει από την κοινή μας παρατήρηση εδώ στην Επιτροπή ότι η Ήπειρός μας αντιμετωπίζει ε, ένα Διεθνέ περιβάλλον ε, με όλο και περισσότερες προκλήσεις που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνο εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη μιλούν με μία φωνή. Είμαι πεπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ευημερήσει σε έναν ε, ε, διασυνδεδεμένο κόσμο εάν αναλάβει το ρόλο μιας, απόλυτης, μιας απόλυτα κυρίαρχης πολιτικής δύναμης. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν συλλογική ηγεσία. Ε, η πολυμερής προσέγγιση βρίσκεται συνεχώς υπό επίθεση και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε νέους συνασπισμούς ε, με χώρες ε, που βλέπουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο με εμά και να έχουμε και ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο. Επανειλημμένα στην Επιτροπή μας έχουμε συζητήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να εξαρτάται από άλλους όσον αφορά την ασφάλειά μας. Και τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια είδαμε κάποια πρόοδο όσον αφορά για παράδειγμα την ε, δημιουργία της ΠΕΣΚΟ, της μόνιμης συνεργασίας. Θα πρέπει όμως να γίνουν περισσότερα για να είμαστε μια σημαντική πολιτική δύναμη στο διεθνές σκηνικό. Υπάρχει ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα. Αποφάσισαν να ε, εστιάσω στα θέματα στρατηγικής σημασίας για την κοινή εξωτερική πολιτική μας ε, και πολιτική ασφάλειας. Γι' αυτό σας παρακαλώ οι τροπολογίες σας να επικεντρωθούν στα κεντρικά θέματα στρατηγικής σημασίας αντί να μπούμε σε λεπτομέρειες που να αφορούν συγκεκριμένες χώρες ή περιφέρειες. Και γιατί το λέω αυτό, διότι έχουμε αρκετές εκθέσεις για διάφορες χώρες στην Επιτροπή μας. Ε, σήμερα ψηφίσαμε πάνω σε κάποιες από αυτές και με όλο το σεβασμό η έκθεση του ΟΗΕ επίσης συζητιέται και ε, υιοθετείται κάθε χρόνο που στη διάρκεια των ετών έχει καταλήξει να είναι μια έκθεση που να ασχολείται με συγκεκριμένες χώρες και συγκρούσεις. Εγώ λοιπόν θέλω να αποφύγω η έκθεση για την ε, ΚΕΠΑ να είναι απλά μια αντιγραφή άλλων εκθέσεων. Τέλος, ε, θα ήθελα να τονίσω ότι ε, θα έχουμε και την ετήσια έκθεση CNSDP για ε, τη Επιτροπή ΣΕΝΤΕ και πολλά θέματα θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε εκείνη την έκθεση και όχι στη δική μα για την ΚΕΠΑ. Προσλέπω στη συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέρφους ε, όπως και πέρσι. Πολύ θα χαρώ να ακούσω τις απόψεις σας πριν την υποβολή τροπολογιών για να έχουμε μια διαρθρωμένη και εστιασμένη συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της ΚΕΠΑ. Περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας πάνω στην έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ομιλητές. Ο κύριος Φλέκενστάιν θέλει να πάρει το λόγο, η κυρία Βαλέρο, ε, ο Στρεβίτσιος, κυρία Γκόμες. Θα ξεκινήσουμε από τον Κνούτ Φλέκενστάιν, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ μπορώ να είμαι σχετικά σύντομος. Καταρχάς, ευχαριστώ θερμά για το γενικά ισορροπημένο σχέδιο έκθεσης που μας έχετε υποβάλει. Όπως είπατε και εσείς, ε, το κείμενο εστιάζει στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και όχι σε συγκεκριμένες χώρες. Μπορώ να σας καθησυχάσω από πλευράς των σοσιαλδημοκρατικών δεν θα λάβετε ε, πολλές τροπολογίες που να έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες χώρες. Ε, συμφωνούμε με τη γενική προσέγγιση. Μία παρατήρηση θα ήθελα να κάνω. Κατά τη γνώμη μου δεν έχετε επικεντρωθεί επαρκώς ε, στα δυνατά σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα σημεία που αναφέρονται στην ε, ήπια ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του soft power. Βάση για αυτήν την ε, ισχύ είναι ο διάλογος. Όποτε είναι δυνατόν ε, με τους γειτόνους μας και άλλους θα πρέπει να επιδιώκουμε τον διάλογο. Και θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το εργαλείο αυτό ε, στα μέσα που έχει στη διάθεσή της η ύπατη εκπρόσωπος. Κατά τα άλλα θα ήθελα να ενισχύσω και την συμβολή των ε, πολιτικών αποστολών όσον αφορά το στρατιωτικό τμήμα. Ε, θα το καλύψει και αυτό η ε, έκθεση. Πάντως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που θέλετε να στείλετε. Είναι λοιπόν σημαντική η έκθεση αυτή για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φλέκενστάιν. Από το, το ECR δεν θέλει να μιλήσει κανείς. Άλτε. Κάτι ακόμη. Ναι, ε, θα με συγχωρήσετε διότι πρέπει να αποχωρήσω. Ε, δεν νόμιζα ότι θα διαρκέσει τόσο η συνεδρίαση. Ζητώ συγγνώμη. Σε ευχαριστώ, Κνούτ. Καλό ταξίδι, Οστρεβίτσιους. Μιλώ εκ μέρους του κ. Φανμπάλεν, που είναι ο σκιώδης ηγητής των φιλελευθέρων. Ζητά συγγνώμη που δεν είναι παρόν σήμερα. Ο κ. Φαν θέλει να σας ευχαριστήσει σας, κύριε Σίγητα, για την με το πολύ καλό προσχέδιο έκθεση. Το βλέπουμε θετικά. Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεισφέρει σε μια αποτελεσματική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι πολλέ προκλήσεις του καιρού μα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί έχουμε ε, προκλήσεις σχετικές με τις, ε, τη δράση της Ρωσίας, τις οποίες πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε ε, αποτελεσματικά. Ο κ. Βαν Μπάλεν λοιπόν θα υποβάλει κάποιες τροπολογίες ε, χωρίς να λιώνει την ουσία του κειμένου. Θα καλύπτουν συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές όπως την κατάσταση στην ε, περιοχή της Ινδίας και του Ειρηνικού. Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία και είναι αισιόδοξο ότι το τελικό κείμενο θα είναι εξαιρετικό και θα είναι έτοιμο μέχρι την Ολομέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος, για τους πράσινους Δεσποίνης Βαλέρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αντικαθιστώ τον συνάδελφο Ταμάς που ε, συνήθως ασχολείται με το θέμα αυτό. Θα είμαι λοιπόν πολύ σύντομη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό Εάν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστος παράγοντας στη διεθνή σκηνή, θα πρέπει να έχουμε φιλόδοξο Φιλόδοξη, αξιόπιστη και κοινή εξωτερική πολιτική που θα πρέπει να συμβαδίζει με ε, οικονομικούς πόρους. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής πολιτική βούληση στα κράτη-μέλη. Επίσης, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, υποχρέωση να στηρίξει τη δημοκρατία και τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα που απορρέει από τις ε, συνθήκες. Σε μερικές φορές όμως βλέπουμε απόλυτη έλλειψη ε, ομοφωνίας ανάμεσα στην στην πολιτική και τελικά στις ε, δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοκρατία και η αρχή του κράτους δικαίου θα πρέπει να τηρούνται. Ανησυχώ όμως όταν μιλάμε με ανθρώπους ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιμένουν η Ένωση να διασφαλίσει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μα θεωρούν όμως απόλυτα αξιόπιστου πια. Θα πρέπει, πιστεύουμε, να υπάρχει καλύτερη ε, σχέση ανάμεσα στους ε, διάφορους τομείς πολιτικής. Έχουμε μια στρατιωτική πολιτική, έχουμε μια πολιτική για τη δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε όμως και πολιτική για τις εξαγωγές όπλων και ε, μερικές φορές ε, αυτές ε, αντιφάσκουν η μία στην άλλη. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που υπόθηκε, ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τις πολιτικές δράσεις. Διότι η κοινή εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφαλείας συμπεριλαμβάνουν την υποχρέωση να, διαχειριζόμαστε κρίσεις Δεν ε, συμπεριλαμβάνει όμως την υποχρέωση διαχείρισης της μετανάστευσης που επίσης είναι πρόβλημα. Δεν ε, θα αναφερθώ αναλυτικά τις ε, τροπολογίε που θα υποβάλουμε θα έχουν όμως να κάνουν με την αξιοπιστία της ευρωπαϊκής πολιτικής και την ε, ενίσχυση της πολιτικής διάσταση ε, σε σχέση με τη στρατιωτική. Thank you, Ms. Ευχαριστώ πολύ, κυρία, κυρία Βαλέρα. Μιλήσατε εκ μέρου του κύριου Μέζεριτ για την Γκουε η κυρία Λόζινγκ. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή. Γενικά, Κάνατε πολλές σωστές παρατηρήσεις. Ναι, πράγματι, η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωση έχει γίνει πιο πολύπλοκη. Πράγματι, πολλοί άνθρωποι ζουν σε πολύ ασταθείς ε, πόλεις και χώρες. Οι χώρες της Δύσης τα τελευταία χρόνια ε, συμπεριφέρονται με τρόπο προτεξιονιστικό και εθνικιστικό. Ενώ χώρες όπως η Κίνα, για παράδειγμα, συνεχίζουν να γίνονται όλο και πιο ισχυρές οικονομικά. Το θέμα είναι τι συμπεράσματα πρέπει να βγάλουμε από όλα αυτά. Σήμερα ήδη το πρωί θέσαμε πολύ σημαντικά ερωτήματα στα πάνελ διότι αναφερθήκαμε στις στρατηγικές για επίλυση των προβλημάτων αυτών με βιώσιμο τρόπο και με σωστές πολιτικές. Πώς ε, θέλει να φέρεται ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, διεθνή σκηνή, τι ρόλο θα μπορέσει να παίξει. Και εμείς από την GUE NGL Πιστεύουμε ότι στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται στρα... στρατηγικές που θα πρέπει που μάλλον αντί για πρόληψη κρίσεων ε, επικεντρώνονται σε στρατιωτικές ε, επεμβάσεις και μεταφέρεται έτσι το βάρος και και καταργούνται οι άλλες δυνατότητες. Ε, γι' αυτό θα υποβάλουμε σχετικές ε, τροπολογίες ε, και θα εκπονήσουμε και μία έκθεση της μειοψηφία. Ιδιαίτερη μας ενδιαφέρει να έχουμε ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα και να βρούμε σωστές πολιτικές λύσεις. και να αναπτυχθούν κατάλληλες στρατηγικές και πολιτικές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, με την ΠΕΣΚΟ έχουμε, πρόβλημα, έχουμε ένα πρόβλημα δημοκρατίας διότι όταν περνάμε από την ομοφωνία στην, ε, στην πλειοψηφία τότε ε, κάποιες χώρες έχουν ε, την δυνατότητα να διαμορφώνουν ε, περισσότερο την εξωτερική πολιτική όσον αφορά τη μόνιμη διαρθωμένη συνεργασία και έτσι από μια ενωμένη Ευρώπη πρέπει να προχωρήσουμε σε μια Ευρώπη που να μπορεί να επηρεάζει τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λούιζινγκ. Σας παρακαλούμε και ε, στην ε, έκθεση ε, για την ΕΠΑ θα σας παρακαλούσαμε να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας, όχι μόνο στο πλαίσιο της δικής μου, πολιτικής, της δικής μου έκθεσης. Η κυρία Κόμες. Είναι ενδιαφέρουσα η έκθεσή σας Πρόεδρε. Διαβάζετε εύκολα. Και αυτό είναι σημαντικό. Τη διάβασα. Έχω έτοιμες τροπολογίες μου. Θα τις λάβετε σύντομα. Νομίζω θα έπρεπε να είμαστε, να είμαστε πιο φιλόδοξοι σε ένα σημείο. Καταλαβαίνω ότι εννοείται ότι έχουμε και την άλλη έκθεση για την πολιτική ασφαλείας και άμυνας, αλλά και αυτή την άσκηση, και αυτή την συγγνώμη, έκθεση θα πρέπει να την τοποθετήσουμε κατά κάποιο τρόπο και στο πλαίσιο της Αμυντικής Ένωσης. Μιλάτε συχνά για την ευρωπαϊκή κυριαρχία και λέτε γι' αυτό χρειαζόμαστε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Ακούγεται λίγο σαν να είναι λόγια του Μακρό, βέβαια, αλλά εκτός αυτού, κατά την άποψή μου, χρειάζεται να πούμε ότι έχουμε ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας. Πρέπει εμείς να μπορούμε να αποφασίζουμε ποιο είναι το συμφέρον μας, τι θα κάνουμε στην παγκόσμια σκηνή και βέβαια να έχουμε και τα μέσα για να υλοποιήσουμε αυτά μας τα σχέδια. Τώρα, σε, τα μέσα, ε, για να υλοποιήσουμε αυτά μας τα σχέδια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέσα τα ίδια, γίνεται μια σύνδεση ανάμεσα στους πόρους και τη μετανάστευση. Ο Σαν, το θέμα, το πρόβλημα της μετανάστευσης να μπορούσε να λυθεί δίνοντας, ρίχνοντας λεφτά στο τραπέζι. Αν οι αναπτυξιακέ οι πολιτικές εξακολουθήσουν να μην δημιουργούν ανάπτυξη, ε, τότε αυτό δεν θα επιτευχθεί, όσα λεφτά και αν ρίξουμε. Και δεν πρόκειται μόνο για τι αναπτυξιακέ πολιτικές, μιλάμε και για την εμπορική πολιτική, για την γεωργική πολιτική κλπ. Χρειάζεται ισχυρέ κοινωνίε των πολιτών, χρειάζεται ε, διαφάνεια, χρειάζεται λογοδοσία, χρειάζεται καλή διακυβέρνηση. Οπότε Όσε επιτροπές και να έχουμε, εμπορίου, ανάπτυξη κλπ. Αν όλα αυτά μεταξύ του δεν είναι δεμένα, δεν δημιουργούν ένα σύνολο συνεκτικό, τότε δεν θα πετύχουμε. Γι' αυτό το λόγο εκεί η ύπατη εκπρόσωπο μπορεί να προσφέρει πολλά. Η ύπατη εκπρόσωπο βέβαια είναι και αντιπρόσωπος της Κομισιόν, έχει δύο ιδιότητε, αλλά θα μπορούσε να ενισχυθεί ο ρόλος της. Επίσης καταλαβαίνουν ότι δεν θέλετε να πούμε να μιλήσουμε για συγκεκριμένες περιστάσεις ή περιπτώσεις. Όμως ίσως θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο ομοί στη γλώσσα μας. Γιατί ε, σε ορισμένες περιοχές στις οποίες η Ευρώπη θα έπρεπε να είναι πιο παρούσα, όπως για παράδειγμα στη Συρία και τη Λιβύη, δεν το καταφέραμε. τι κάναμε, το μόνο που προσφέραμε ήταν ανθρωπιστική βοήθεια, το ελάχιστο δηλαδή. Και γιατί δεν τα καταφέραμε, γιατί τα κράτη-μέλη ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ε, ευχαριστώ, Άννα Γκόμες. Δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα επιθυμούσαν να πάρουν το λόγο. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ από το τμήμα στρατηγικής ε, πολιτικής από την Κομισιόν αν θα ήθελε να πάρει το λόγο. Πού είναι? Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά με βρίσκει σύμφωνο αυτό το σχέδιο έκθεσης που πραγματικά προσπαθεί να δει σε γενικές γραμμές την όλη εικόνα. Πραγματικά είναι μάλλον ζωφερή η εικόνα. Ε, υπάρχει θέμα αστάθειας. Από την άλλη πλευρά διαπιστώνουμε επίσης ότι υπάρχουν ορισμένοι τομείς όπου επιτελείται πρόοδος σε ό,τι αφορά τη συνδεσιμότητα, τη μετανάστευση, ε, και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που δείχνουν ότι όταν πραγματικά καταβάλουμε προσπάθεια μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι ε, και το θέμα των, του επίπεδου των προσδοκιών σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Αυτό τι σημαίνει για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά θα πρέπει να δράσουμε όλοι μαζί και είναι ενδιαφέρον να, δούμε πόσοι από τους όρους που χρησιμοποιήθηκαν σήμερα, ας πούμε ευρωπαϊκή κυριαρχία, αυτονομία, αναφέρονται όλο και περισσότερο στους Ευρωπαίους ηγέτες και τη συζήτηση που γίνεται για αυτό το θέμα. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να έχουμε συνείδηση το πόσο ευάλωτοι είμαστε σε ορισμένους τομείς. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, τα συμφέροντά μας, να έχουμε σταθερές αξίες, αλλά και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά όταν επιλέγουμε τις δεσμεύσεις μας με τους εταίρους μας. Αυτό είναι που αποκαλούμε ο ευρωπαϊκός δρόμος, ο ευρωπαϊκός τρόπος. Και εδώ συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που έχουν σχέση με την άμυνα, ε, αλλά και στοιχεία που ήταν γνωστά στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένως θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας ορισμένους τομείς, να χαλαρώσουμε σε άλλους. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας στην Ευρώπη, το θέμα είναι πώς μπορούμε να προφυλάξουμε καλύτερα τα συμφέροντά μας, πώς θα πρέπει να κινηθούμε σε επίπεδο περιφερειακό και πώς θα μπορέσουμε ε, να ε, προφυλάξουμε ε, όλες τις πτυχές, όλες τις πλευρές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα μπορούσαμε να επιλέξουμε καλύτερα τις στρατηγικές μας και να ε, συμφωνήσουμε ένα νέο προϋπολογισμό στο ε, πολιετές ε, πλαίσιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε στρατηγικές κατευθύνσεις όταν υιοθετηθεί αυτή η πρόταση. Πραγματικά περιμένουμε να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και να συνεργαστούμε με την Επιτροπή ΑΦΕΤ και είμαι στην διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση. Merci bien. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντεφάν. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τη νέα γραφή, γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο ε, να είμαστε ε, μεγαλειώδεις στα μεγάλα, αλλά και πιο σκληροί στα σκληρά και πιο μαλακοί στα μαλακά. Καταπληκτικά πράγματα είναι αυτά που ακούσαμε. Συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε. Με μεγάλη υπομονησία περιμένω τις τροπολογίες σας. Ελπίζω να έχουμε μια καλή συνεργασία με τους κοιόδης, να βρούμε συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Ντέφαν. Ε, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 11 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί και θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή στις 21 Νοεμβρίου σε αυτή την Επιτροπή και τον Δεκέμβριο στην Ολομέρεια. Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα τώρα να δώσω την ε, σκητάλη στην Αντιπρόεδρο. Ποιος, ποιος θα προεδρεύσει. Α, Ντουμπάφκα, εσύ θα προεδρεύσεις. Έχουμε το 24 και το 25. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε διευρυμένο προεδρείο στις 6 παρατέταρτο. Ας προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τη συνάντηση, τη συνεδρίαση αυτή στις 6 παρατέταρτο. Ας συνεχίσουμε, όπως είπε ο Πρόεδρός μας. Έχουμε τώρα μια κοινή συζήτηση των σημείων 24 και 25. Συμφωνία υπομορφή ανταλλαγή επιστολών μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με την τροποποίηση των πρωτοκόλων 1 και 4 τη Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών του αφενό και του Βασιλείου του Μαρόκου αφετέρου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 Και για τις δύο γνωμοδοτήσεις είναι συντάκτης ο κύριος Βίστησεν. Χωρίς πολλά πολλά, να του δώσω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Φτάνουμε στη γνωμοδότηση που θα υποβάλουμε σε σχέση με την απόφαση ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ε, συμφωνία με το Μαρόκο. Ε, στην απόφαση αυτή υποβλήθηκαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τροποποίηση της εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Σαχάρας για να είναι νόμιμη η συμφωνία. Πρόκειται για έκθεση της ΙΝΤΑ. Η ΑΦΕΤ ζήτησε να γνωμοδοτήσει Λόγω όμως χρονικού περιορισμού από ό,τι κατάλαβα από πλευρά ε, της Επιτροπής Ίντα αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Οπότε εμείς απλά γνωμοδοτούμε στην γνωμοδότηση της Ίντα πάνω στη Συμφωνία Υπομορφή Ανταλλαγής Επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής ε, Κοινότητας ε, και του Βασιλείου του Μαρόκου. Τα δύο βασικά κομμάτια της απόφασης είναι καταρχάς η αξιολόγηση του οικονομικού όφελους προς τον πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας και το άλλο που αφορά ιδιαίτερα την ΑΦΕΤ είναι η διαβούλευση ε, του τοπικού πληθυσμού. Και κατά τη γνώμη μου, σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωθεί η δική μας γνωμοδότηση και γι' αυτό έχω υποβάλει σχετικά σύντομες γνωμοδοτήσεις ε, που θα σταλούν στην Επιτροπή Ίντα που ε, επαναλαμβάνουν τα σημαντικά θέματα. Για παράδειγμα, ε, τις προσπάθειες του ΟΗΕ για μια λύση στη Δυτική Σαχάρα. Αναφέρομαι όμως και στην ΕΙΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, συμμόρφωση με την απόφαση του δικαστηρίου στα δύο θέματα που προανέφερα. Ξέρω ότι είναι καυτό το θέμα αυτό, είναι επίμαχο θέμα. Αυτή τη στιγμή όμως η δική μας δουλειά είναι να εξετάσουμε αυτές ε, τις δύο απαιτήσεις ε, της απόφασης του δικαστηρίου και η ομάδα ECR ζητάει και ανταλλαγή απόψεων με τον ε, ειδικό απεσταλμένο ε, για την ε, Δυτική Σαχάρα γενικά. Καλό όμως τους συναδέρφους να υπερψηφίσουν αυτήν την έκθεση που είναι τεχνικής φύσης και όσον αφορά τα πολιτικά ζητήματα και το καθεστώ ε, τη ε, Δυτική Σαχάρα, να τα συζητήσουμε αυτά σε άλλο πλαίσιο. Αυτά λοιπόν είναι όσα έχω να πω για τι νομοδοτήσει αυτέ. Ε, προσβλέπω στη συνεργασία με του σκιώδεις εισηγητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και του δικού μου βοηθού για τη δουλειά που έχουν κάνει πάνω στο θέμα αυτό. Πολύ ευχαρίστω θα ακούσω τι παρατηρήσει των συναδέρφων. Ευχαριστώ κύριε Βίστησεν. Όπω είπατε, επί τη ουσία αρμόδια είναι η Επιτροπή ΙΝΤΑ. Λόγω όμως της συμφωνίας του θέματος, λόγω της σημασίας του θέματος, αποφασίσαμε και, να, εμείς να υποβαλούμε γνωμοδότηση. Έχω κάποιους συναδέλφους εδώ που θέλουν να πάρουν το λόγο. Καταρχάς ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συζητάμε ένα σημαντικό θέμα που άπτεται των σχέσεων με το Μαρόκο. να υπογραμμίσω μια ακόμα φορά τη σημασία του Μαρόκου ως προνομίου εταίρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο σε διμέρες επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό το επιβέβαιωσε μία ακόμα φορά πρόσφατα η Επιτροπή ΧΑΝ, που πήγε στο Ραμπάτ το Σεπτέμβρη. ο Επίτροπος Χάν, συγγνώμη, όχι η Επιτροπή Χάν, ε, ο οποίος ε, ε, συζήτησε και με τον Υπουργό Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκου είπε ότι θέλει να γυρίσει σελίδα μετά από αρκετά χρόνια εντάσεων και λίγο αργότερα μέσα στο 2018 ο Υπουργός Εξωτερικών του Μαρόκου θα είναι εδώ, θα έρθει εδώ στην Επιτροπή μας να μας μιλήσει. Η έκθεση αυτή ε, φτάνει λοιπόν στην πιο σωστή στιγμή, είναι πολύ επίκαιρη. Το θέμα των επαρχιών του Νότου ήταν πάντοτε περίπλοκο. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να, να αναγνωρίσουμε ότι ε, μια, οι δικές μας συστάσεις δεν θα, βρουν, δεν θα δώσουν λύση στο πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να στηρίξουμε μια να στηλέξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για να επιληθεί το πρόβλημα στο μέλλον. Δεν θα πρέπει να ξαναξεκινήσουμε ε, μια λεκτική διαμάχη. Το πρώτο προσχέδιο του κ. Βίστησεν είναι πολύ καλό, λαμβάνει υπόψη τις παλιότερες συζητήσεις που είχαμε για το θέμα αυτό. Το σημερινό κείμενο είναι καλό σημείο αφετηρία. γιατί αναφέρει ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωση δεν έχει αλλάξει ό,τι αφορά τι επαρχίες του Νότου και εξακολουθούμε να στηρίζουμε τη διαδικασία του ΟΗΕ. Οι έρευνε που έχουν γίνει έχουν αποδείξει ότι οι περιοχές αυτές θα ωφελούν το αν συμπεριλαμβάνονταν στη συμφωνία. Χρειάζονται οικονομική ανάπτυξη, έχουν δικαίωμα να αναπτυχθούν και γι' αυτό το λόγο έχουν δικαίωμα πιο έντονων σχέσεων, πιο στενών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόρριψη αυτών θα αποτελούσε και ένα χτύπημα στις σχέσεις μας, στις σχέσεις μας με το Μαρόκο, αλλά και μια μετακίνηση του παραγωγικού ιστού από αυτές τις ε, περιοχές του Νότιου Μαρόκου στον υπόλοιπη χώρα. Αυτή η κατάσταση άλλωστε θα ήταν και παράλογη. Το βλέπουμε ήδη. Είναι μια κατάσταση που δεν βοηθάει κανέναν. Οπότε πιο λογικό θα ήταν να δημιουργηθεί μια νομική βάση, πραγματική και απτή, και να μην επιτρέψουμε μια, ένα νομικό κενό. Βέβαια, ε, αρμόδια είναι η Επιτροπή Ίντα που θα συζητηθεί και το θέμα της συχνηλασιμότητας των προϊόντων. Θα πρέπει να συζητήσουμε επίσης το πώς θα, τη σήμανση θα τίθεται πάνω σε αυτά τα προϊόντα. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση πάντως. Θα συνεργαστούμε πολύ καλά με τον κύριο Βίστησεν, είμαι σίγουρος, και με τους άλλους και ηγητές. Ελπίζω όμως να εστιάσουμε στο, στην ουσία και να μην καταστεί αυτή η έκθεση μια έκθεση για το Μαρόκο και για τη συνολική περιοχή της Βορειάς Αφρικής. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέντα. Ξέρετε ότι ο κύριος Αλώνης δεν είναι δυστυχώ σήμερα εδώ. Ας συνεχίσουμε με την κυρία Ντεβαλέρο εξ ονόματος των Πρασίνων. Α, και δύο. Α, πρώτο Κλάους, πρώτο Κλάους, γιατί πρέπει να φύγει. Παρακαλώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνουμε τη διάκριση. Δεν είναι αλήθεια αυτό που υπόθηκε επανειλημμένα ότι πρόκειται για τις νότιες περιφέρειες του Μαρόκου. Είναι παράνομη κατεχόμενη περιοχή. Αυτό έχει διαπιστώσει και ο ΟΗΕ και Ε, τρομάζομαι αυτό που ακούω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα προσπαθήσει να βρει ε, τρόπους να παρακάμψει την απόφαση του δικαστηρίου. Το έχει ακόνει αυτό με τον εξή τρόπο. Έχει γίνει ανταλλαγή πληθυσμών στην Δυτική Σαχάρα χωρίς ε, να ε, ερωτηθούν οι άνθρωποι αυτοί ε, και χωρίς να ερωτηθούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι φυλακισμένοι που υφίστανται βασανιστήρια τα οποία θέτουν σε κίνδυνο και τη ζωή τους. Η Επιτροπή Ίντα επισκέφθηκε τη Δυτική Σαχάρα, θέλησε να συνομιλήσει με μη κυβερνητική οργάνωση. Και η αστυνομία εμπόδισε τέτοιες ε, συνομιλίες. Η αστυνομία συνόδευε συνεχώς την αποστολή μας ε, και εμπόδισε οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση και συνομιλία. Ο πρέσβης ε, παρενέβη για να προσπαθήσει να βελτιώσει το κλίμα, αλλά νομίζω ότι απέτυχε. Βλέπουμε ε, ε, κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμένα μου φαίνεται τρομερό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρεί τον εαυτό της κοινότητα αξιών παραβιάζει ψηφίσματα του ΟΗΕ και παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Σα uh, Σας ευχαριστώ κύριε Μπούχνερ. Υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει να πάρει το λόγο. Η κυρία Βαλέρο, αλλά νομίζω πρώτα... Ε, να ακούσουμε όχι τους ε, φιλελεύθερους, αλλά ε, την ε, αντιπροσωπεία για την Σαχάρα. Κύριε Γιάννα Σέντερ, ε, είναι καλή αυτή η έκθεση, ισορροπημένη, η έκθεση του κύριου Βίστησεν. Η... Περιγράφει τις δράσεις της Κομισιόν μετά την απόφαση του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχολιάζει σωστά. Αναγνωρίζω ότι πολλοί δεν συμφωνούν, αλλά δεν θα λύσουμε εμείς το πρόβλημα της ε, Δυτικής Σαχάρας. Αυτό που πρέπει είναι να μην δημιουργούμε σοβαρά προβλήματα, να μην επιδεινώσουμε τα προβλήματα ούτε των επαρχιών του Νότου, ούτε της κυβέρνησης του Μαρόκου, κυβέρνηση του Μαρόκου που βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια δύσκολη συγκυρία, ως ε, ιδιαίτερος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζεται στενά μαζί μας και στην καταπολέμηση τρομοκρατίας και στην ε, χαλιναγώγηση της ε, μετανάστευσης μέσω νομιμοποίησης μεταναστών που ζουν στο Μαρόκο. Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι το έργο της, μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε μας αρέσει είτε όχι, ε, έχει σεβαστεί την αποφάση του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι που διαφωνούν ζητούν μια καινούργια απογραφή και ένα καινούργιο δημοψήφισμα, κάτι που δεν μας αφορά όμως εμάς. Ε, η αλήθεια είναι ότι έχουν κληθεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το Πολυσάριο να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Το, πολυσάριο, το μέτωπο Πολυσάριο δεν συμφώνησε για τους δικούς του λόγους ε, για να συζητήσουν. Εμείς, λαμβάνοντας υπόψη ε, εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη το σύνολο της πραγματικότητας, όχι μόνο ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Οπότε πολύ σωστά αντιμετωπίζει το ζήτημα ο κύριος Βίστισεν και ζητώ να υπερψηφιστεί. Ευχαριστώ, Παρακαλώ, Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω σχετικά. Ε, παρακαλώ λοιπόν να φορέσετε τα ακουστικά σας. όπω και ο συνάδελφο Κλάου, θα ήθελα να αποστασιοποιηθώ από το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε τη συμφωνία αυτή. Έχω εξετάσει και την ε, έκθεση της κυρίας Λαλόντ και αναφέρονται οι μη αυτόνομες περιοχές αντί για τις νότιες περιοχές όπως ε, αναφέρθηκε πριν. Δεν μιλάμε όμως ούτε για νότιες περιφέρειες ούτε για μη αυτόνομες. Μιλάμε για κατεχόμενα εδάφη. Τα δύο τρίτα αυτών είναι κατεχόμενα. Έχει γίνει ανταλλαγή πληθυσμού ώστε η πλειοψηφία Αυτόν που μένουν εκεί να είναι μαροκινή ε, μαροκινοί ε, έπικοι. Ενώ ο ντόπιο πληθυσμό ε, στην πλειοψηφία του ζει σε καταβλισμούς στην Αλγερία. Αυτή λοιπόν η συμφωνία που προσπαθούμε να περάσουμε από εδώ πέρα αντίκειται στην απόφαση του δικαστηρίου. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτά συνάδουν με την απόφαση του δικαστηρίου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παρακάμψουμε την, ε, τις συνέπειες της απόφασης αυτής. Ήταν απόλυτα σαφές ότι η Δυτική Σαχάρα δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία με το Μαρόκο. Το Μαρόκο ε, δεν ε, έχει καμία αξίωση να πουλά προϊόντα από την Δυτική Σαχάρα. Επίσης, ε, δεν αναγνωρίζουμε το Πολυσάριο ως εκπροσώπους ε, του, ε, της Δυτικής Σαχάρας. Αυτό όμως ε, το κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ η Σουηδία να έχει πει ότι δεν αναγνωρίζει το Πολυσάριο ως θεμητό εκπρόσωπο της Δυτικής Σαχάρας. Ταυτόχρονα λέμε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τις ε, δράσεις ε, του ΟΗΕ για να βρεθεί η λύση στην ε, διαμάχη αυτή για τη Δυτική Σαχάρα και θα πρέπει να βασίζεται αυτό στην αυτοδιάθεση των Σαχράουι. Γιατί λοιπόν δεν τους επιτρέπουμε να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα που τους υποσχέθηκαν πριν τόσα χρόνια. Αντί λοιπόν να στηρίζουμε τον ΟΗΕ στη δουλειά του, κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Υπονομεύουμε τις προσπάθειες του ΟΗΕ να πετύχει λύση στη διαμάχη αυτή. Όσον αφορά την διαδικασία διαβούλευσης, 112 οργανισμοί προσκλήθηκαν. Ενώ 94 οργανισμοί δεν έλαβαν την πρόσκληση ή αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Ε, το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, μίλησε με ανθρώπους στη Δυτική Σαχάρα, μίλησε μαζί με εκπροσώπους είτε στο Ραμπάτ είτε στις Βρυξέλλες. Αυτό όμως δεν είναι σωστή διαβούλευση ε, εγκαταλείπουμε στη μοίρα τους, ε, τους ανθρώπους της ε, Δυτικής Σαχάρας και αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Το θέμα δεν είναι ότι πρέπει εμείς να βρούμε λύση για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά το Πολυσάριο εκπροσωπεί τους ανθρώπους αυτούς και αυτοί θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, όχι οι έπικοι κατεχομένων εδαφών. Ευχαριστώ. Okay. Thank you, Mrs. Ωραία. Ευχαριστώ, κύριο Βαλερό. Ο κύριος Πίκατ. Όπως γνωρίστηκε, ξεκίνησε, ξεκίνησαν διαβουλεύσεις το Συμβούλιο ζήτησε να ζητηθεί η άποψη του πληθυσμού του Δυτικής Σαχάρας για αυτή τη συμφωνία και είναι πολύ ενδιαφέρον για μας πώς πήγαν αυτές οι διαβουλεύσεις. Κύριε Πίκατ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, εκπροσωπώ την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Δίπλα μου είναι πρόσωπος της Επιτροπής. Και δεν θέλω να μιλήσω για το θέμα των ε, διαπραγματεύσεων, των διαβουλεύσεων, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να πω ότι μας βρίσκει σύμφωνο το σχέδιο κειμένου